Ε, θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Πριν παράσουμε στο επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη, έχω μία πληροφορία να σας πω. Η κυρία Άννα Μιράντα με ενημέρωσε ότι παρετείται από την Ευρωβουλή από τις 10 Ιουλίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3 του εσωτερικού κανονισμού, το Κοινοβούλιο καταγράφει αυτό το γεγονός και βλέπει και σημειώνει ότι υπάρχει ε, μια κενή έδρα και ενημερώνει τις, σχετική, τις σχετικές αρμόδιες αρχές. Και το πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.